Παρακαλώ καθίστε. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας και φτάσαμε στον τέταρτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ε, εκλέξουμε, να κληρώσουμε μάλλον ένα νέο ψηφολέκτη που θα αντικαταστήσει την κυρία Ντότς. Αν έχετε την καλοσύνη να μας φέρετε εδώ την κάλπη για να κληρώσουμε έναν αντικαταστάτη της κυρίας Ντότς. Η κυρία Λάρα Κόμη, παρακαλώ, αντικαθιστά την κυρία Ντότς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κόμι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε λοιπόν στον τέταρτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσω ότι με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού κατά τον τέταρτο γύρο υποψήφιοι είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι κατά τον τρίτο γύρο συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Δηλαδή οι κύριοι Πιτέλα και Ταγιάννη. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω να μοιραστούν ε, τα ψηφοδέλτια παρακαλώ τους ε, ψηφολέκτες ε, να κάτσουν στη θέση τους. Κυρία Κόμη, πρέπει να κάτσε στη θέση της κυρία Ντότς, στην θέση παριθμών 3 που βλέπετε θα σας δείξουν, ε, θα σας δείξουν ακριβώς που πρέπει να πάτε. Ο κύριος Χέκμαρκ, ε, όταν έχει κάτσει ο κύριος Χέκμαρκ, τότε πια ε, είμαι και σίγουρος ότι όλα πάνε καλά. Ο κύριος Χέκμαρκ λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχει κάτσει στη θέση του κατόπιν τούτου. Κυρίες και κύριοι, έλαβαν τη θέση τους όλοι οι ψηφολέκτες. Πολύ ωραία. Άρχεται λοιπόν ο τέταρτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας. Meine Damen und Herren, alle ihre Stimme abgegeben. Κυρίες και κύριοι, ψηφίσατε όλοι. Από ό,τι βλέπω όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτησή μου. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Μήπως ε, επιθυμεί κάποιος ε, να ψηφίσει τώρα που δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Τα περιμένω, προφανώς και τα περιμένω μέχρι να ψηφίσετε όλοι. So, letzter Aufruf. Λοιπόν, για τελευταία φορά ερωτώ, ε, ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Αν ψηφίσατε όλοι, κλείνει ο γύρος, ο τελευταίος γύρος. Παρακαλώ οι ψηφολέκτες ε, να μεταβούν στην αίθουσα R11 και θα ακούσετε το κουδούνι για να επανέλθετε στην Ολομέλεια ή αν θέλετε μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες όπου θα προβάλλετε το σχετικό μήνυμα προβλέπω ότι το αποτέλεσμα θα το έχουμε μεταξύ 9 η ώρα και 9 και 4. Μέχρι τότε λύεται η συνεδρίαση.